είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για την κατάσταση στο Σουδάν. Να δώσω απευθείας το λόγο στον Υπουργό κ. Κούρκουλα. Παρακαλώ. President, honorable members, Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι μας λυπεί ιδιαίτερα η αναφορά ενός, ε, να, ε, ατυχήματος με ferry ε, που 120 άτομα έχασαν τη ζωή τους στον νυχτά του Νότια Σουδάν. Ε, συλληπούμεθα τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Αυτό το τραγικό περιστατικό ε, προσθέτει ένα αριθμό νεκρών στον ήδη μεγάλο αριθμό θυμάτων ε, στο Νότιο Σουδάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαίτερα από την χειροτέρευση της ανθρωπιστικής κατάστασης και από αναφορές ε, μεγάλης κλίμακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, 10.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 400.000 ε, έχουν ε, εγκαταλείψει τις αιστείες τους στο Νότιο Σουδάν, ενώ περίπου 15.000 έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Πέρα από αυτό, αυτή η κρίση ε, ενέχει τον κίνδυνο να επηρεάσει μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή που ήδη ε, ε, χαρακτηρίζεται από βία φτώχεια και ανασφάλεια. Αυτό που συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εξακολουθούμε να ε, θεωρούμε ότι είναι μέλημά μας να υποστηρίξουμε τις διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες να λήξει η βία και καλούμε να ανεβρεθεί μια λύση με πολιτικές διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν στους ηγέτες του Νοτιού Σουδάν να λύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά και δημοκρατικά. Μαζί με την διεθνή κοινότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί, προσπάθησε να προλάβει την κρίση και ε, έτσι ώστε ε, να μην καταλήξει σε εμφύλιο πόλεμο και σε χάος. Έχουμε εκφράσει την πλήρη υποστήριξή μας στην ICAT στην ε, ε, Διεθνή Αρχή Ανάπτυξης ε, Διαμεσολάβησης προκειμένου να κηρυχθεί ανακοχή και να τεθούν οι βάσεις για μια πολιτική δημοκρατική λύση. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σχολιάσω την έκθεση της κυρίας Ντεκάιζερ που υιοθετήθηκε πέρσι το Δεκέμβρη που υπογράμμισε τις προκλήσεις ανάπτυξης ε, ε, οικοδόμησης ε, του κράτους στην, στο Νότιο Σουδάν. Η IGAT είναι αξιέπαινη διότι διαμεσολαβεί ανάμεσα στις δυνάμεις του Νοτιού Σουδάν και ζητούμε από, όλους τις, από όλους τους εμπλεκόμενους να προσπαθήσουν να ζητήσουν λύση πριν να είναι πολύ αργά προκειμένου να αποφευθεί ο εμφύλιος πόλεμος. Η, η τη της Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπος ε, της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ε, έχει ζητήσει να ε, κηρυχθεί ανακοχή και να δοθεί πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια. Η χρήση της ε, βίας ε, δεν θα πετύχει τίποτα. Η, πρόσφατη ιστορία μας, διδά, το έχει διδάξει. Η αντιπρόεδρος κυρία έχει υπογραμμίσει ότι μια άμεση ανακοχή ε, με αποτελεσματική παρακολούθησή της θα πρέπει να συμφωνηθεί το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να γλιτώσει, γλιτώσει ο λαός του Νοτιού Σουδάν από ε, περαιτέρω βάσανα. Ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορέσει να επιτευχθεί σύντομα και ότι ε, μια αξιόπιστη ανακοχή θα υπογραφεί σύντομα όπως ο ε, αντιπρόσωπος του τύπου του Πρόεδρου Σαλβακίρ έδειξε να εννοεί. Η κυρία Άστον έχει ενθαρρύνει τα μέρη να δημιουργήσουν συνθήκες για έναν ε, ειρηνικό πολιτικό διάλογο που θα, περιλαμβάνει, που θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των πολιτικών ηγετών που αυτή τη στιγμή κρατούνται στην πρωτεύουσα Γιούμπα έχει καλέσει τα δύο μέρη να αποφύγουν δημόσιες δηλώσεις που θα ε, μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους οπαδούς τους να προχωρήσουν σε περαιτέρω βίες επιθέσεις. Ε, ο, όλοι όσοι ενθαρρύνουν τη βία καθυστερούν την επιτυχία της αναγκοχής, παρεμποδίζουν την πολιτική διαδικασία, ιδιαίτερα στις προσπάθειες ε, μεσολάβησης της ΆΙΚΑΤ και ε, φρενάρουν την ε, πολιτική διευθέτηση του θέματος. Αυτά τα μέρη ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πράξεις τους θα έχουν συνέπειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια αποφασιστική διπλωματική προσπάθεια έτσι ώστε να δοθεί τέλος στη διαμάχη η ε, ειδική εκπρόσωπος, ο ειδικό εκπρόσωπος Αλεξάνδερ Ρόντος ε, για το κέρας Αφρικής ε, βρίσκεται στην περιοχή από τις 25 Δεκεμβρίου και αδιάκοπα ε, βρίσκεται σε επαφή με τους βασικούς παίκτες στο νότιο Ιράν και σε όλη την περιοχή έτσι ώστε να στηρίξει την οικοδόμηση μιας ε, συνένεσης για, υπέρ των προσπαθειών της ΆΙΚΑΤ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έχει προσφερθεί να υποστηρίξει και πολιτικά και οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Είναι σημαντικό ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη πίσω από την IGAT και ε, να υποστηρίξει αυτή τη ε, διαδικασία. Μα ανησυχούν ιδιαίτερα αναφορές παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα τα μέρη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αυτουργή συστηματικών και στοχευμένων ενεργειών παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα δώσουν λόγο η προστασία των ε, πολιτών θα πρέπει να, να, να επιτευχθεί. Ε, καλωσορίζουμε την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης ε, για την σύσταση επιτροπής που θα ερευνήσει ε, καταγγελίες ε, περί παραβίασης του ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, καθώς επίσης και τις βασικές αιτίες και τους παράγοντες που οδήγησαν στη βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Επιτροπή αυτή να ξεκινήσει το έργο της το συντομότερο. Επίσης υποστηρίζουμε ε, την συνεχιζόμενη ενίσχυση της αποστολής του ΟΗΕ στο Σουδάν έτσι ώστε να μπορέσει να ε, προστατεύσει τους ε, πολίτες, τους αμάχους. Η, η, το γραφείο του ΕΚΟ και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και είμαστε έτοιμοι να ε, απομακρύνουμε ε, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης καθώς επίσης και να βοηθήσουμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αντιπροσωπεία στη Γιούμπα. Εξακολουθούμε να δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όσοι χρειάζονται και ήδη από τις 23 Δεκεμβρίου η Επίτροπος ανακοίνωσε 50 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική δράση προκειμένου να καλυφθούν βασικές ανάγκες, πόσιμο νερό, τρόφιμα, προστασία κλπ. Σήμερα, μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δώσει περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια τα έτη 2013-2014. Τελειώνω λέγοντας ότι και επαναλαμβάνοντας ότι ε, πέρα από τις πολλές ε, ζωές που έχουν καταστραφεί, χαθεί, η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν ε, ενέχει τον κίνδυνο ε, να αποσταθεροποιήσει όλη την ε, περιοχή. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί. Όλοι οι ε, παγκόσμιοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Θα πρέπει να ε, δεσμευτούν τα μέρη, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ξεκινήσουν διάλογο. Είναι σημαντικό και επίγον το κόστος ε, του να μην συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι πολύ ψηλό. Το τίμημα θα είναι πολύ σοβαρό για τους πολίτες του ε, Νότιου Σουδάν. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα λαό που ε, πολέμησε ε, στεναρά για την ανεξαρτησία του. Θα πρέπει όλοι μας να παραμείνουμε ονομένοι πίσω από τις προσπάθειες της ΆΙΚΑΤ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να μην φυστεί ε, προσπαθειών προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους ομιλητές εξ ονόματων των πολιτικών ομάδων. Ε, ο κύριος πρέτα για το ΕΛΚ για ε, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Το Δεκέμβριο του 2013 το κοινοβούλιο μας, θα το θυμάστε άλλωστε, ενέκρινε την έκθεση της κυρίας Δεκάιζερ. Έξερα την έκθεση όπου αναφέρθηκαν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για τον Νότιο Σουδάν. Δυστυχώς, λίγες μέρες μετά η... ξεκίνησε η εμπόλεμη σύραξη μεταξύ των στρατευμάτων της κυβέρνησης και των ε, αντιφρονόντων στα πλαίσια των ε, ομάδων του πρώην Αντιπροέδρου με καταστροφικές συνέπειες στην Επιτροπή τη δική μας. Συχνά αναφέρονται και συζητιόνται οι πολιτικές αστάθειες στη χώρα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να ομολογήσω ότι ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα καταλήγαμε στη σημερινή κατάσταση. Ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει ε, διχασμός της χώρας και να δημιουργηθεί μια κατάσταση που θα υπάρχει ε, ανατολικό και δυτικό Νότιο Σουδάν. Έχουν χαθεί πολλές ζωές και διαπιστώνουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά ιδιαίτερως έντονα τις τελευταίες εβδομάδες. Κάθε θετικό σημάδι το οποίο λαμβάνουμε από την περιοχή αυτή θα έπρεπε να το καλωσορίσουμε. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου το είπε και συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι η Αφρικανική Ένωση ε, θέλει να συστήσει μια επιτροπή διερευνητική και ο πρόεδρος Αλβακία αλλά και ο Ριέτ Μασά θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους από πολιτικής άποψης γιατί και οι δύο ευθύνονται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να τις αποτρέψουν αυτές τις παραβιάσεις ε, εις βάρος των αμάχων. Θα πρέπει να, να ε, σταματήσει η διαμάχες και να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον Νότιο Σουδάν, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και την εκκίνηση μια διαδικασία εθνικής συμβιλίωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ των Σοσιαλιστών, η κυρία Ντεκεζέρ για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη λύπη μου έμαθα τον αριθμό των θυμάτων ε, στο Νότιο Σουδάν Πρόκειται για τραγωδία και συμφωνώ απολύτως ε, ε, ότι πρέπει να συλληπιθούμε τον λαό του Σουδάν, στον οποίο αξίζουν σίγουρα πολύ καλύτερα πράγματα. θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιήθηκε επί τόπου και θα πρέπει να πω ότι τρεις από τους υπαλλήλους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μείνει σήμερα στην Τζούμπα και κάνουν εξαιρετικό έργο. Σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Ένωση, η διεθνής κοινότητα και η Τρόικα ε, την οποία αποτελούν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία, ε, δραστηριοποιήθηκαν αμέσως και έφτασαν επιτόπου στο Νότιο Σιδάν μόλις ανακήρυξε την ανεξαρτησία του όταν ακόμα δεν υπήρχε ούτε καν μία δομή που θα μπορούσε να βοηθήσει το κράτος από τις εκθέσεις που ψηφίσαμε υπάρχει και η έκθεση του Δεκεμβρίου η οποία ήδη επεσήμανε ότι επιθυμούμε τη σταθερότητα αυτού του νέου κράτους και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ελλείμματα σε θέματα δημοκρατίας, σε θέματα παιδείας υπάρχουν ε, εθνοτικές διαμάχες, ε, παραστρατιωτικές ομάδες και όλα αυτά τα πράγματα ε, μας έδειχναν ότι ελοχεύει ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος κυρίως με τις γείτονες χώρες και την ε, από βορρά ε, απειλή. Αλλά ε, δεν περιμέναμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή η οποία συνέβη. Από το 2011 έως το 2013 διαθέσαμε 830 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη αυτής της χώρας. Έχουμε προβλέψει 1.300.000 μέχρι το 16 και θα πρέπει να προβλέψουμε και περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, ο IGAD ε, το υποστηρίζεται από πλευρά σήμερα, υποστηρίζουμε την Αφροκανική Ένωση και πρέπει να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε και θα πρέπει κυρία Πρόεδρε και με αυτό ολοκληρώνω εν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, Ένωσης και του IGAD να συζητήσουμε το θέμα της δημοκρατία δημοκρατίας σε μια χώρα στην οποία πρεσβεύει η διαφθορά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια τέτοια ευάλωτη χώρα έρμεο των κινδύνων τους οποίους βιώνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρος, ο κύριος Λουί Μισελ για δύο λεπτά. Ναι. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κρίση του Νοτιού Σουδάν προέρχεται από πολλές πηγές όπως αναφέρθηκε ε, εθνοτικοί διχασμοί, το γεγονός ότι υπάρχει η διαμάχη για το πετρέλαιο επίσης, ε, κάποιες στρατηγικές ε, αντιπαλότητες και φυσικά και οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Η εξαιρετική έκθεση της κυρίας Δεκεζέρ είχε ήδη επισημάνει τους κινδύνους και τα ευάλωτα σημεία που έχει μια τέτοια χώρα η οποία είναι ε, στη διαδικασία της γέννησής της. Πέραν λοιπόν από το γεγονός ότι πλήττεται ο λαός ε, του Νοτιού Σουδάν που έχουμε πολλούς εκτοπισμένους και πρόσφυγες, η κρίση που βιώνει το Νότιο Σουδάν απειλεί σαφώς και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ουγγάντα, η λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ε, όλες αυτές οι χώρες ε, κινδυνεύουν ακριβώς ε, γιατί και οι ίδιες είναι σε ευάλωτη θέση και πολύ μακρινό είναι ένα μέλλον στο οποίο πραγματικά θα μπορούμε να σκεφτούμε μια λύση. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και στον πρόεδρο Σαρβάκη και στον αντιπρόεδρό του, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο αντίπολός του, ότι δεν θα πρέπει να καταφύγουν στη βία και στην εθνοτική διαμάχη η οποία έχει ξεκινήσει και είναι εξελίξη. Θα θέλαμε να ζητήσουμε άμεση κατάπαυση πυρών, να υπάρχει πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, να υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικές οι οποίες θα προκύψουν καταρχάς από την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ ε, την επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τον Νότιο Σουδάν, η οποία δεν έχει προσπάθειες προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα και ε, βοηθά την ΆΙΓΑΤ, η οποία προσπαθεί να ε, επαναφέρει την τάξη στη χώρα είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Σουδάν. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προβλέψουμε και μία ε, παράταση της εντολής ε, του Αλεξάνδρου Ροντόρφ, του ειδικού εκπροσώπου για την Αφρική, ε, ο οποίος μετέβει επιτόπου και έχει αποκαταστήσει τις τακτικές επαφές μεταξύ του Προέδρου του Νοτιού Σουδάν και της ευρύτερης περιοχής. Το να μην παραταθεί η θητεία του σημαίνει ότι δεν θέλουμε να δεσμευτούμε επαρκώς στο θέμα αυτό. Βεβαίω Βεβαίως ε, επιμένουμε ότι όποια παραβίαση υπάρχει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, ό,τι πρέπει να γίνει για να προστατευτεί ο άμαχος πληθυσμός θα πρέπει να γίνει, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί να απο... προκειμένου να αποφύγουμε εμφύλια σύραξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντουρά δεν είναι στην αίθουσα. για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, είναι ε, απίστευτο που πριν από ένα μήνα είχαμε αναγνωρίσει ε, την πρόοδο του Νοτιού Σουδάν ε, προς την ανεξαρτησία του και τους ενθαρρύναμε να προβούν σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να εδραιώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες το Νότιο Σουδάν βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού με συνδυασμό πολιτικών αντιζηλιών ε, αντικυβερνητικών ανησυχιών για εξαιτίας ε, της διανομής των κερδών από το πετρέλαιο και εντάσεις, φυλετικές εντάσεις. Ε, υπάρχει ε, μια αντιπαλότητα μεταξύ δύο ανθρώπων, του πρόεδρου με τον, τον αντιπρόεδρο, που έχει κοστίσει ε, σε χιλιάδες άτομα τη ζωή του. Πολύ περισσότερο μετά το τελευταίο ατύχημα που, που έχασαν τη ζωή του 200 άτομα και ε, έδειξε το τι κάνουν για να ξεφύγουν από, τον, από την εμπόλεμη κατάσταση. Το κράτος αυτό είναι ιδιαίτερα εύθραυστο, ε, είναι νέα δημοκρατία, λείπουν οι θεσμοί, οπότε ε, κανείς δεν ξέρει πόσο, πόση πίεση και αίμα θα μπορέσει να αντέξει πριν διαλυθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για το λαό, αλλά και πολύ επικίνδυνο και αποσταθεροποιητικό για όλη την περιοχή του κέρατος Αφρικής. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που στο παρελθόν έχει υποστηρίξει τον Νότιο Σουδάν πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις για την ανακοχή. Καλωσορίζω τις εργασίες του ειδικού εκπροσώπου στο κέρας της Αφρικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις προσπάθειες της ε, Αφρικανικής Ένωσης και της ICAT. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης τεχνικά και οικονομικά τους πρόσφυγες ε, αν οι διαπραγματεύσει αποτύχουν και η κατάσταση εξελιχθεί σε φίλιο πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει ακόμα και στρατιωτική επέμβαση ε, παράλληλα με την ανθρωπιστική της δράση. Και ορίζω την πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης να δημιουργήσει, ε, να συστήσει επιτροπή, διερευνητική επιτροπή το Νότιο Σουδάν ε, έχει ε, πετρέλαιο, ε, μπορεί να βαστεί σε αυτό, αλλά δεν μπορεί να αντέξει ένα φίλο πόλεμο. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το σταματήσουμε. Για την ΚΟΥΕ τώρα, η κυρία Λούζινγκ, 1,5 λεπτό. Όταν από πλευρά της Ευρώπης εξετάζουμε τις βίες συγκρούσεις ε, στην Αφρική μιλάμε συχνά για εθνοτικέ αιτίε. Η σημερινή αυτή η διαμάχη προέρχεται από τέτοιους αιτίε. Αυτό ισχυρίζονται ε, ο τύπος και εδώ στο Κοινοβούλιο αρκετές φωνές. Αυτό δεν αφαιρεί την οικονομική κατάσταση που είναι καταστροφική η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν χαρακτηρίζεται από πολλαπλές συγκρούσεις σε ένα κράτος που εξαρτάται πλέον από την υποστήριξή μας. Οι βασικοί παράγοντες ε, συγκαταλέγονται σε διαφορετικές ε, εθνότητες, αλλά αυτό είναι τυχαίο ίσως. Είναι μεγάλη η γεωστρατηγική τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα. Και αυτό, αυτές οι συγκρούσεις ενισχύουν τα συμφέροντα των ελίτ. Παρά τον πλούτο σε πετρέλαιο, τον πλούτο της χώρας, ο πληθυσμός είναι σε μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Είναι κοινική η κατάσταση. Η διάβρυνση της σύγκρουσης στην ε, περιφέρεια ανησυχεί την εθνική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτό ζητώ την ε, χορήγηση όπλων άμεσα στην περιφέρεια, στην περιοχή αυτή. Και θα πρέπει λοιπόν έτσι η χώρα να επιλύσει τα πραγματικά της προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Ε, η κυρία Γκαμπριέλη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Πρόκειται για μια χώρα η οποία ήδη βρίσκεται σε αδύναμη θέση λόγω των πρόσφατων σειράξεων, αλλά η εμφύλια διαμάχη έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για την περιοχή. Θα πρέπει καταρχάς ε, με κάθε τρόπο να αποφύγουμε τον πόλεμο και κυρίως να μην λάβει περισσότερο εθνοτικές διαστάσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι γυναίκες και τα παιδιά του Νότιου Σουδάν αναγκάζονται να υπόκεινται σε όλες αυτές τις ε, ταλαιπωρίες ανεξάρτητα από το σε ποια εθνοτική ομάδα ανήκουν. Θα πρέπει να προστατεύσουμε κυρίως τους αμάχους και αυτή θα πρέπει να είναι η βασική αποστολή της κυβέρνησης, ακόμα και αυτούς που θεωρούν από εναστάτες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική λύση μέσω των όπλων. Η λύση θα πρέπει να είναι δημοκρατική και πολιτική. Χωρίς κατάπαυση πυρών δεν θα μπορέσει να υπάρξει καμία ε, λύση για τις δύο πλευρές. Η ομάδα της ΆΙΚΑΤ θα πρέπει λοιπόν να επιμείνει στη διαδικασία αυτή και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διαμεσολαβητές. Και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσει και η Αφρικανική Ένωση για να μπορέσει να ε, βοηθήσει ώστε να μην μεταδοθεί η κρίση στις υπόλοιπες χώρες της ε, Αφρικής, του κέρατος της Αφρικής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανάγκε των αμάχων είναι κατεπίγουσες, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν και κατάλληλε δημοκρατικές δομές. Θα πρέπει η διαδικασία μετάβασης να είναι διάφανη και ακόμα και για τους πόρους. Και θα πρέπει η ε, διεθνής κοινότητα να μην χάσει αυτό το στόχο από τα μάτια της. Δεν θα πρέπει οι πιο ε, στερημένες περιοχές του κόσμου να είναι και οι πιο εφήμερες δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Λάστρα για 1,5 λεπτό. Το εξ Αυτοεξονόματο ε, παραπάνω από τριών εκατομμυρίων ε, ατόμων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια και ε, των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τι αιστείε του κάνει έκκληση να σταματήσουν αμέσω οι επιθέσει εναντίον αμάχων και να ξεκινήσει ένα διάλογο και να δημιουργηθεί ένα οδικό χάρτη προ την ειρήνη. Ε, το Νότιο Σουδάν ήταν σε πόλεμο με το, βόρειο, ε, με το Σουδάν ήδη για αρκετό καιρό κάτι που δημιούργησε ε, πολλά, προκάλεσε πολλά θύματα αυτή τη στιγμή το αίμα ρέει και η οι φτωχοί και πεινασμένοι πολίτες ζητούν ένα κράτος δημοκρατικό και ειρηνικό ο δρόμος προς την ειρήνη απαιτεί την ε, ε, δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου. Ε, η ειρήνη θα περάσει μέσα από την, ε, το, το τέλος της ε, βίας και από τον αφοπλισμό. Θα πρέπει όσοι παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα να λογοδοτήσουν. Το ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο δυναμικός. Θα πρέπει να ε, βοηθήσει την Αφρικανική Ένωση και στις προσπάθειές της να αποφευχθεί η διεύρυνση και η γενίκευση του πολέμου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Ευχαριστώ. Το να περάσουμε τώρα στη διαδικασία του Catch Α, συγγνώμη. Η κυρία Γκόμες για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Τρία χρόνια μετά την ανεξαρτησία η βία και τα βάσανα επέστρεψαν στο Νότιο Σουδάν. Η ανθρωπιστική καταστροφή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τις τοπικές ε, ε, και τις περιφερειακές οργανώσεις. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την ΑΕΓΑΤ και προκειμένου να κηρυχθεί ανακοχή να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι και να ε, ενθαρρύνουμε τους πολιτικούς ηγέτες να εγκαταλείψουν την βία. Ενώ ταυτόχρονα όσοι ε, προέβησαν σε αδικήματα θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Η διεθνής κοινότητα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια σε, ε, στις δομές ε, του Νοτιού Σουδάν και στη οικοδόμηση ενός κράτους. Η στρατηγική μας αυτή κινδυνεύει. Ε, αυτή τη στιγμή ε, οι, οι πολιτικές ελίτ ε, υποθάλπουν ε, φιλετικές διαφορές και δημιουργούν διαφθορά. Θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση να βοηθεί να συμμετάσχει, να αναλάβει την ευθύνη να πείσει τους πολιτικούς ηγέτες και να εξασφαλίσει ε, μια μεταβατική κυβέρνηση μέχρι το 2015 στο πλαίσιο μιας ε, ειρηνευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, φυλές και θα αποφύγει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει το Νότιο Σουδάν, στο Νότιο Σουδάν να σταματήσει η εσωτερική διαμάχη και να μην χρησιμοποιηθεί από το καθεστώς του Αλμπασίρ από το Βορρά και από άλλες ε, δυνάμεις της περιοχής. Γι' αυτό τον λόγο υποστηρίζω την ανανέωση της ε, θητείας του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΚΕΑ της Αφρικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΗ. Ο κύριος Στίερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Νότιο Σουδάν ξεκίνησε και έπεσε σε ένα νέο φαύλο κύκλο της βίας ε, το Δεκέμβριο του περσινού έτους μετά από τη σύγκρουση μεταξύ Πρόεδρου και Αντιπρόεδρου. Δυστυχώς ε, στο Νότιο Σουδάν δεν κατάφερε να διατηρήσει μετά την ανεξαρτησία του την ε, ειρήνη και αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπάρξουν νέες αποχρώσεις, ε, για παράδειγμα και οι εθνικές ε, αποχρώσεις πέρα από τις πολιτικές ε, προτιμήσεις. Έχουν προσθεθεί πολλοί πρόσφυγες, τους ήδη αριθμούς πρόσφυγες και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Η χώρα έχει καταλήξει παρόλα αυτά όμως σε ένα διέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν να τα επιλύσουμε αυτά τα θέματα για να μην τιμωρούνται αθώοι άνθρωποι άμαχοι. Ευχαριστώ. Μπαζέσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Νότιο Σουδάν ενδεχομένω να θέσει σε κίνδυνο και την σταθερότητα όλη τη περιφέρεια. Δύο χρόνια μετά την ανεξαρτησία, διαπιστώνουμε πόσο ασθενεί είναι οι θεσμοί στη χώρα δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την επικράτη της χώρας και ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλοί άμαχοι κινδυνεύουν από την βία της ε, κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. οι νεκροί, άριθμοι και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Και ο αριθμός των ε, θυμάτων θα αυξηθεί. Δυστυχώς η ανθρωπιστική κατάσταση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την ε, πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν οι συγκρούσεις, ύστερα θα πρέπει να υπάρξει πρόοδο σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο Νότιο Σουδάν. Ευχαριστώ κύριε Ορόλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για το πιο νέο κράτος του κόσμου και η κατάσταση λοιπόν είναι ιδιαίτερα ευάλωτη από την ανεξαρτησία και μετά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί μια νέα ελπίδα στη χώρα αυτή και να δοθεί όλη η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια για την ε, ειρήνευση. Φαίνεται ότι οι τοπικές οργανώσεις έχουν κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος τους για την ε, επιτεύξη της ειρήνης. Την, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχα την ευκαιρία να συζητήσω τα θέματα αυτά με τον πρώην Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, τον κύριο Μπούντερικ. Και κατέστησα σαφέ ότι στο Σουδάν είναι απαραίτητο είναι απαραίτητη η δημοκρατική τεχνογνωσία, το πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα, πώς θα πρέπει να δρά η κυβέρνηση. Είναι καλό το γεγονός ότι η ίδια οργάνωση έχει κάνει σημαντική δουλειά στη χώρα αυτή και σε άλλες χώρες άλλωστε. Επίσης και η ηλική βοήθεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να λάβουμε την ευθύνη μας και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να αποστέλουμε μια αποστολή για την διαχείριση της κρίσης στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κρόμπεργκερ. Σας ευχαριστώ θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να κάνουμε πολλά περισσότερα σε ό,τι αφορά την κρίση αυτή. Χρειάζεται κατεπηγόντως βοήθεια και η Ευρώπη θα πρέπει να την παράσχει. Θα θέλαμε να καλέσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμουν στην ε, ε, αποστολή του ΟΗΕ με αστυνομικέ και στρατιωτικέ δυνάμει. Και βλέπουμε διάφορες δομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπω ε, η ΚΕΠΑ. Θα πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία προγραμματισμού για μια επόμενη αποστολή μετά την ε, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να, κινητοποιηθούμε για τον αφοπλισμό και καλούμε την ύπατη εκπρόσωπο να υποστηρίξει την διακυβερνητική αρχή και τις ε, ε, διαπραγματεύσεις προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα παροχή βοήθειας και μια μεσολάβηση που θα διευκολύνει την όλη κατάσταση. Χρειαζόμαστε πραγματικά καλύτερο συντονισμό, καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της, ε, των ΗΠΑ, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ κύριε Βεργιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η λύση που μας ε, υποβάλλεται δεν ε, ε, δημιουργεί καμία αμφιβολία για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο Νότιο Σουδάν. Για άλλη μια φορά έχουμε ε, χρήση για πολιτικούς σκοπιούς ε, των διαφόρων ομάδων που ζουν στην περιοχή. Χειραγώγηση από πλευράς μας. Και αυτό είναι στις πηγές των όσων συμβαίνουν. Σήμερα ε, γίνεται συμμαχία με τον Αλμπαζίρ ε, για τη διαχείριση των πετρελαίων. Υπάρχει ο δικτάτορας του Βορρά και εκεί έχουν ε, συγκεντρωθεί όλο και περισσότερα μέρη του πληθυσμού. Υπάρχει η στρατιωτική προδοσία όπως λέγεται για τους πολιτικούς υπευθύνους. Έχουν φυλακιστεί οι άνθρωποι του πρώην αντιπροέδρου, άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, υπάρχουν χιλιάδες πρόσφυγες και θα πρέπει ε, να δούμε τι ακριβώς τίμημα πρέπει να πληρώσει ο λαός του Σουδάν για να μπορέσει να υπάρξει ειρήνη. Χρειαζόμαστε μια πολιτική λύση και για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει να κάνει κάτι για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Υπουργό κύριο Κούρκουλα. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση στο Νότιο Σουδάν ξεκίνησε πριν από λιγότερο από ένα μήνα. Ε, κατά βάση υπάρχει, γιατί είναι μια πολιτική διαμάχη, η οποία κλιμακώθηκε σε ε, βία. Για να σταματήσουμε να αποφύγουμε μια ακόμα καταστροφή στην περιοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, αυτή η κρίση δεν θα ε, λυθεί με περισσότερη βία. Δεύτερον, η ΆΙΓΑΤ ε, αρκετά γρήγορα έθεσε τον εαυτό της στο επίκεντρο των ε, προσπαθειών διαμεσολάβησης. Αυτό θα πρέπει και να επενεθεί και να υποστηριχτεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει όλες τις διεθνείς και περιφερειακές προσπάθειες να ευθυγραμμιστούν και να υποστηρίξουν τις ε, προσπάθειες διαμεσολάβησης της ΆΙΚΑΤ και αποθαρρύνει οποιαδήποτε εξωτερική επέμβαση που θα μπορούσε να εντείνει τις ε, εσωτερικές διαμάχες του Νότιου Σουδάν. Τρίτον, θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ε, όλη, οποιαδήποτε βία κατά μάχων θα πρέπει επίσης να σταματήσει και οι υπεύθυνοι ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν. Τέταρτον, Παρόλο ότι η διένεξη ξεκίνησε πριν από λιγότερο από ένα μήνα, οι αιτίε είναι πολύ πιο βαθίε Και η επίλυση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω ενός σταθερού διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές που θα έχει ως στόχο την, ε, ε, να οδηγηθούμε σε μια συμφιλίωση, εθνική συμφιλίωση που θα περιλαμβάνει όλες τις πλευρές. Δεύτερον, όλες οι πλευρές θα πρέπει να επιτρέψουν ε, αμέσως ε, και χωρίς όρους στην ανθρωπιστική βοήθεια έτσι ώστε να βοηθούν χιλιάδες ε, Σουδανοί, νοτισουδανοί υπήκοοι που είναι τα πραγματικά θύματα της βίας. Ε, αν η διαμάχη συνεχιστεί θα αυξηθεί ο κίνδυνος να μετατραπεί σε φίλιο πόλεμο. όλο και περισσότεροι ε, άνθρωποι θα ε, χάνουν τη ζωή τους ή θα αναγκαστούνται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και αυτοί που προσπαθούν να μείνουν στο περιθώριο θα αναγκαστούν και αυτοί να συμμετάσχουν στην, ε, να πάρουν μέρος ε, στην διαμάχη. Θα πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών και σίγουρα αν αποτύχουμε θα χρειαστεί να λογοδοτήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος Ολοκληρώνεται η συζήτηση και ψηφοφορία αύριο 5η 16 Ιανουαρίου. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κοινή συζήτηση, εμπερικές συμφωνίες με το Μεξικό και τη Χιλή. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή.